Καλό καθίστε. So, ich darf Sie Θα ήθελα λοιπόν ε, να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε σήμερα μία συζήτηση με δύο κύρια σημεία. Πρώτον, νέες μορφές εργασίας. Κάτι που έχουμε χωρίσει σε δύο γύρους. Μία ώρα θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ε, διότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ και δεύτερον, θα ασχοληθούμε με την ε, εποπτεία και παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών για άτομα με αναπηρίες ε, ως μόνιμο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Καταρχάς, ε, θέλω να σας ε, μιλήσω για κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση. Θα συμπροεδρεύσω μαζί με τον συνάδελφο Άντριαν Σόλομον, που είναι πρόεδρος ε, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας. Εγώ λέγομαι Τόμας Χέντελ, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μοιραστούμε λοιπόν το καθήκον της Προεδρίας σήμερα το απόγευμα. Ε, τη διαδικασία τη γνωρίζετε. Όποιος έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ να συμπληρώσει τη σχετική κάρτα και να μας την παραδώσει. Δύο λεπτά ε, χρόνος ε, ομιλίας προβλέπεται για τον καθένα. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ, αλλά μπορώ να σας καθησυχάσω ότι στο Κοινοβούλιο συχνά έχουμε μόνο ένα λεπτό χρόνο ομιλίας. Θα προχωρήσουμε ως εξής. Τρεις εθνικοί βουλευτές θα πάρουν το λόγο. Προτού να ξαναδώσουμε το λόγο σε έναν ευρωβουλευτή ή μία ευρωβουλευτή. Έτσι θα έχουμε την σωστή εναλλαγή και σωστή συμμεταχή των συναδέρφων από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τμήμα των εργασιών μας. Ε, θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε γρήγορα, διότι 6 και 10 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο της ε, συζήτησης και να προχωρήσουμε στο δεύτερο τμήμα για να κλείσουμε στις 7 η ώρα, για να μην πεθάνετε από την πείνα και για να πάμε για το δείπνο. Αυτά λοιπόν, ο Άντριον Σόλομον θα μας κάνει μια εισαγωγή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την συνεδρίασή μας, κύριε Σέρκα. Είμαι ο κύριος Σέρκας Κόζε και η κυρία Ράντα Βαλτσόβδαν. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε να συμμετάσχετε σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ανάδυση νέων μορφών απασχόλησης, κύριε Κόζε, αντιπροσωπεύουν τις αξίες που εκπορεύονται από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Εργασιακών Δικαιωμάτων. Διαπιστώνουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ψηφιοποίηση, η ρομποτοποίηση είναι ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις συνάμα για το εργασιακό δυναμικό, για την ποιότητα της εργασίας και των συνθηκών εργασίας, για τις εργασιακές σχέσεις, για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και την εργασιακή ζωή. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές τροποποιήσεις της αγοράς εργασίας μετά από την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή δεν αποτελούν μόνο ευκαιρίες διαφοροποίησης της αγοράς εργασίας και, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν και θέσεις απασχόλησης κυρίως για τους νέους. Ωστόσο, συνοδεύονται από πολύ ισχυρέ ανησυχίες για τις συνθήκες εργασίας, για το ύψος του εισοδήματος και για την κατανομή των εισοδημάτων, των εσόδων. Υπ' αυτή την έννοια τα κράτη-μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν συμβάσεις εργασίας μη τυπικές να τηρούνται και να γίνονται σεβαστά. Θα πρέπει τα κρατημέλη να λάβουν μέτρα έτσι ώστε να έχουμε διαφάνεια και ε, προβλεψιμότητα στις συνθήκες εργασίας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να δώσω το λόγο στον πρώτο συνομιλητή, στον κύριο Κόσε, μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εισαγωγικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να μιλήσω για την εργασιακή ζωή στο μέλλον. Η εργασία και οι συνθήκες εργασίας ε, παίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Είναι κάτι που επηρεάζει τη ζωή μας, το πώς νιώθουμε, πώς ζούμε, ακόμα και το πόσο ζούμε. Έχουμε τώρα μία αγορά εργασίας ε, που έχει αλλάξει ριζικά. Έχουμε δει νέες μορφές απασχόλησης ε, και έχουμε επίσης ψηφιοποίηση η οποία επηρεάζει τη ζωή μας, πώς δουλεύουμε, ακόμη και το πώς ε, κάνουμε τα ψώνια μας. Έχει αλλάξει η δομή της αγοράς εργασίας τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε νέα τεχνολογία, ε, νέα ψηφιακά συστήματα και έχουμε αυτοματοποιήσει πολλές διαδικασίες. Ταυτόχρονα έχουμε την οικονομία του διαμοιρασμού. Έτσι λοιπόν έχουμε και ε, εργασιακές και φορολογικές προκλήσεις η ευελιξία αυξάνεται και έχουμε τις πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας σε, σε τομείς όπου εργάζονται κυρίως γυναίκες, όπως για παράδειγμα ο τομέας ε, των ε, ξενοδοχείων ή της εστίασης. Επίσης ε, βλέπουμε πολλούς νέους ανθρώπους ή ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό που εργάζονται στους τομείς αυτούς. Ο εργοδότης ε, θεωρείται ότι μπορεί να μειώσει τον χρόνο εργασίας ε, για τους εργαζομένους, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια ερωτήματα στο πλαίσιο αυτό. Πώς μπορούμε να έχουμε πιο ευέλικτες μορφές εργασίες, ε, πώς, μπορούμε να πώς είναι δυνατόν να έχουν όλη πρόσβαση σε, στην εργασία. Σε πολλές χώρες έχουμε ακούσια μερική απασχόληση. Και βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ε, παρότι εργάζονται. Πώς λοιπόν μπορούμε να εγγυηθούμε αξιοπρεπή εργασία για τους εργαζομένους και πώς μπορούμε να φροντίσουμε οι ε, μορφές απασχόλησης αυτή τη στιγμή να μην εγκατασταθούν από ακόμα χειρότερες. Έχουμε λοιπόν ψηφιοποίηση, ρομποτοποίηση, ε, τεχνητή νοημοσύνη και οι αλλαγές αυτές έχουν ε, οδηγήσει και σε αλλαγή της αντίληψής μας ε, για την εργασία. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε την ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να βρούμε καινοτομίε για να βελτιώσουμε τη ζωή για εκατομμύρια ανθρώπων, να χρησιμοποιήσουμε νέε τεχνολογίε για να έχουμε πιο καθαρέ και πιο βιώσιμε ε, ε κοινωνίε και καλέ συνθήκε εργασία για όλου. Θα ήθελα να ε, παραθέσω τα λόγια του Γιώραν Γιώρανσον από το Πόρκ που είπε ότι δεν φοβάμαι τη νέα τεχνολογία, φοβάμαι την παλαιά. Και αναμφίβολα θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις τα επόμενα χρόνια, θα ακούσουμε νέες ιδίες, θα απορρίψουμε παλιές θεωρίες. Αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων ιδεών και την ε, δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για διαβίου μάθηση. Θα χρειάζονται συχνά επανεκπαίδευση οι άνθρωποι σε μια αγορά εργασίας που θα εξελίσσεται συνεχώ. Επίση, χρειαζόμαστε βελτιωμένο κοινωνικό διάλογο. Η αγορά ε αναφέρεται συχνά ως, ε, ως παιχνίδι μηδενικού ε, αθροίσματος. Δηλαδή, αν κερδίσει ο ένα, θα χάσει ο άλλο. Αλλά αυτό είναι λάθο, γιατί ένα ισχυρό κοινωνικό διάλογο συχνά βοηθεί σε ε, καλύτερε συνθήκε για του εργαζομένου και περισσότερη σταθερότητα και ε, μεγαλύτερη παραγωγικότητα για του εργοδότε. Α έχουμε λοιπόν μια κατάσταση win-win από την οποία κερδίζουν όλοι. Τρίτον, χρειαζόμαστε και κοινωνική πρόνοια και ε, ασφάλεια. Θα πρέπει να επενδύσουμε στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, να έχουμε καλύτερη φροντίδα ε, παιδιών για να μπορέσουν να εισέλθουν ε, περισσότεροι στην αγορά εργασία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία κάτι που έχει θετικά αποτελέσματα σε σχεδόν όλους τους τομείς. Στην ανάπτυξη, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Είναι λοιπόν δυνατά όλα αυτά. Ναι. Θα χρειαστούν πολλές ε, προσπάθειες, συνεργασία και πολιτική βούληση. απολύτω. Προσβλέπω στο να θέσουμε μαζί τη βάση για μια εργασιακή ζωή όπου όλοι να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Je suis été euh, donné la parole. Θα ήθελα τώρα να δώσω την κυρία Καμάτσοβα, πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ε, κυρία Μαξοβά, παρακαλώ. Děkuji, Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, έχω ετοιμάσει μία σύντομη παρουσίαση στα αγγλικά, θα μιλήσω όμως τσέχικα. Στην Τσεχία, όπως και σε όλη την Ευρώπη, βλέπουμε την ανάπτυξη νέων ειδών εργασίας. Και αυτό δεν σημαίνει ότι οι θέσεις απασχόλησης εξαφανίζονται, αλλά περιμένουμε έναν σημαντικό μετασχηματισμό όπου θα συνδυάζονται διαφόρων ειδών δραστηριότητες. Για παράδειγμα, θα συνδυάζεται η ανθρώπινη εργασία ε, με ε, τα μηχανήματα. Αυτό προσφέρει ευκαιρίες στους εργαζομένους και στους εργοδότες. Ε, μπορούμε όλοι να υποφεληθούμε από την πρόοδο της τεχνολογίας. Ευελιξία και απασχόληση για τις ομάδες που αυτή τη στιγμή έχουν δύσκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, ε, για γονείς, ε, για φροντιστές, και για ανθρώπους σε, σε μειονεκτικές περιοχές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε εναλλακτικές λύσεις καθώς και νομική διευκόλυνση ώστε να πετύχουμε με ομαδικό πνεύμα ε, καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές ε, στις οποίες ε, εμπίπτουν και η χρήση της ρομποτοποίησης. Θα πρέπει κυρίως ε, να παρέχουμε την κατάλληλη ευελιξία για τον συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, όμως και κάποιοι κίνδυνοι, κάποιες θέσεις απασχόλησης χάνονται. και ε, επίσης ε, υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες για ανθρώπους με χαμηλές δεξιότητες ε, ή με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. Η, οργάνωση της εργασίας αλλάζει, η ασφάλεια για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Με τις νέες μορφές εργασίας εργοδότες αναμένεται να ενδιαφερθούν λιγότερο για την μετεκπαίδευση των εργαζομένων και αυξάνεται το κόστος εκπαίδευσης. Επίσης υπάρχουν κίνδυνοι για ιδιαίτερες ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν λιγότερες ψηφιακές δεξιότητες και χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης στο μέλλον οι θέσεις απασχόλησης ε, θα είναι όλο και πιο επισφαλείς. Και γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η προστασία των εργαζομένων, καθώς ε, και η κοινωνική ασφάλιση και η ιατρική περίθαλψη. Επίσης, οι ε, τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής μπορεί να δημιουργήσουν άγχος και να έχουν αρνητικές συνέπειες στους εργαζομένους. Στο μέλλον ε, θα αναμένεται να γίνουμε όλο και πιο παραγωγικοί, διότι μέσα στα επόμενα 20 χρόνια το 10% των ε, θέσεων απασχόλησης ε, αναμένεται να απολεθούν λόγω της αυτοματοποίησης και θα επηρεαστεί το 35% των θέσεων απασχόλησης. Μέχρι το 2029 αναμένεται να χαθούν ε, συνολικά 420.000 θέσεις απασχόλησης και να αλλάξουν ε, θέση απασχόλησης σε 1,4 εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτά τα στοιχεία συνδέονται ε, λιγότερο με ε, τους ανθρώπους με υψηλές ε, τεχνικές ε, και ψηφιακές δεξιότητες. Εκεί περιμένουμε πιο σταθερή κατάσταση. Επίσης, στο μέλλον θα χρειάζονται όλο και περισσότεροι χειριστές μηχανών και η ψηφιοποίηση θα παίξει σημαντικό ρόλο. Ενώ αναμένεται αύξηση στον τομέα των υπηρεσιών ο πληθυσμός ε, γυράσκει και θα πρέπει να δούμε τι μορφές απασχόλησης ε, μπορούν να ε, χρησιμοποιηθούν για τους ανθρώπους αυτούς. Έχουμε επίσης την οικονομία του διαμοιρασμού, έχουμε άλλες μορφές υπηρεσιών και η περιφερειακή κατανομή των ε, θέσεων απασχόλησης ε, δεν ε, θα είναι πολύ ίση. Έχουμε και διάφορες πλατφόρμες όπως είναι το Airbnb και άλλες. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες αλλάζουν τις μορφές απασχόλησης Ε, παρέχουν περισσότερη ευελιξία. Μπορεί κανείς να ε, πετύχει τη συμμετοχή ανθρώπων από διάφορες περιοχές. Τέλος, ε, τι μπορούμε να περιμένουμε. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλους τους τομείς της οικονομίας θα πρέπει να εξετάσουμε το καθεστώς του, τον ορισμό του παρόχου υπηρεσιών και επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, σωστούς κανόνες για την ε, ασφάλιση υγείας και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην μονοπολούν ελάχιστες πλατφόρμες σε την όλη ε, αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μεξόβα. Τώρα θα τα πω στα ρουμάνικα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ανταλλαγή απόψεων και θα δώσω το λόγο στην κυρία Αγγέλοβα Σβέτλοβα από την, ε, Βουλγαρία και νομίζω ότι είναι μέλος της Επιτροπής ε, Κοινωνικών Υποθέσεων από το ΕΛΚ. Κυρία Αγγέλοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, αλλάζει με δυναμικό τρόπο η αγορά εργασίας και επομένως μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Εμείς στη Βουλγαρία έχουμε σημαντική οικονομική ανάπτυξη, η αγορά εργασίας βελτιώνεται, ωστόσο η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην προσφορά ε, και τη ζήτηση σχετικά με το εργατικό δυναμικό εξακολουθεί να υπάρχει, να δημιουργεί πρόβλημα. Ε, προτείνονται βεβαίως κάποιοι μηχανισμοί έτσι ώστε να μειωθούν αυτές οι ανισορροπίες και κάθε χρόνο ε, η ε, κυβέρνηση, η χώρα ε, λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθούν οι γνώσεις και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Άλλωστε αυτό είναι και το σλόγγαν. Αυτό που θέλουμε είναι εργατικό δυναμικό το οποίο να έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Στα πλαίσια του ε, επιχειρησιακού προγράμματος ξεκινήσαμε πολλές ε, δράσεις ε, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και των μονοπρόσωπων επιχειρήσεων. Ε, είναι σημαντικό να ε, συμπεριληφθούν σε όλα τα προγράμματα ε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ανεργία ή δεν έχουν γνώσεις και μέσω της απόκτησης γνώσεων θα μπορέσουν να βρουν θέση εργασίας. Το 2019 θα είναι μια μεγάλη χρονιά για τις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ε, θα ε, συγχρηματοδοτήσουν κατά 50% γιατί το υπόλοιπο 50% το χρηματοδοτεί ο δημόσιος προϋπολογισμός. Θα χρηματοδοτήσουν, λέω, ε, κατάρτιση και εκπαίδευση που θα βοηθήσει για τις νέες μορφές απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. για τα όσα μας είπατε, αγαπητή κυρία Αγγέλοβα. Ντέμπορα Σεραγιάννη από την Ιταλία. Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης της Βουλής από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, in Italia, Ευχαριστώ. Στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια εμείς ε, κάναμε μια σημαντική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας που οδεύει προς την κατεύθυνση που οι δύο εισηγητέ ανέφεραν προηγουμένως. Δηλαδή κάναμε επένδυση λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και την κρίση ε, όσον αφορά σημαντικές αρχές ευελιξίας. Ε, και τώρα έφτασε και η στιγμή να περάσουμε από την προηγούμενη αντίληψη της ποσότητας στην τωρινή αντίληψη Τη ποιότητα. Μιλάμε για σχέσει εργασία ορισμένου χρόνου ή νέε σχέσει εργασία, για νέε μορφές εργασίας που ακόμα δεν ε, αναγνωρίζονται σωστά σε ένα σύστημα το οποίο εντωμεταξύ δεν έχει προσαρμοστεί στις τεχνολογικές και άλλες ε, ε, ε, καινοτομίες. Ε, αυτή είναι και η ερώτηση μάλιστα που θέλω να κάνω στους εισηγητές στα πλαίσια της παρούσης συζητήσεως. Η αντίστοιχη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτίθεται να προωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοβουλίες που θα αφορούν όλες τις χώρες μέλη, ας πούμε όσον αφορά κάποια αποζημίωση ανεργίας που θα είναι ενιαία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που θα διευκόλυνε και την μεταφορά καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μελών. Δύο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθενται να ε, ε, επενδύσουν σε ένα σημαντικό και συνολικό πρόγραμμα ε, επανεκπαίδευσης εργαζομένων που κινδυνεύουν να μείνουν έξω από το νέο σύστημα εργασίας έτσι όπως διαμορφώνεται. Στην Ιταλία έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία αυτή, αλλά θα θέλαμε κάποιο κίνητρο και από την Κομισιόν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ από την ε, Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν πρόφερα σωστά το όνομά σα, λέει ο Πρόεδρος. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, όταν μιλούμε για την κατάσταση στην Ευρώπη και στην Κύπρο σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και την κατάσταση των εργαζομένων, το πρώτο που χρειάζεται να προσδιορίσουμε είναι ότι αυτό που τα καθορίζει είναι η κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης εκδοχής του καπιταλισμού τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στις χώρες μέλη. Η ρυθμισμένη εργασία μέσα από συλλογικέ συμβάσεις απασχόλησης στοχοποιείται ως υπέτεια για την ακαψία της οικονομίας. Ο θεσμός της σύνδεσης των μισθών με τον πληθωρισμό οι μισθολογικές κλίμακες, οι προσαυξήσεις, ο κατώτατος μισθός θεωρούνται αυτοματισμοί που διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η σταθερή η μόνιμη απασχόληση θεωρείται εμπόδιο στην προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων. Τα δημόσια συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης θεωρούνται υπέρμετρο βάρο στα δημόσια οικονομικά με τη λύση να δίνεται στην κατεύθυνση της μείωσης των συντάξεων, στην επέκταση ή κατάργηση των ορίων συνταξιοδότησης και την προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι οργανισμοί που είναι κρατική ιδιοκτησία θεωρούνται ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και ότι αποτελούν βάρος για τα δημόσια οικονομικά. Η διασφάλιση από το κράτος βασικών αγαθών για όλους τους πολίτες, υγεία, παιδεία, στέγαση, όπως και τα καθολικά επιδοματά, θεωρούνται ως μηχανισμοί που στρεβλώνουν τον υγιή και ανώθευτον ανταγωνισμό και εμποδίζουν την ελεύθερη λειτουργία της οικονομίας. Έτσι, παρά το γεγονό ότι οι εργασιακέ σχέσει και τα θέματα κοινωνική πολιτική με βάση τη συνθήκη τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν εθνικέ αρμοδιότητε, στην πράξη μέσα από τι διατάξει του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και άλλε παραμέτρου, το νεοφιλελεύθερο μοντέλο επιβάλλεται σε όλες τις χώρες ε, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία της απορρίθμισης ήταν πολύ πιο εντονή και βίαιη στις χώρες που μπήκαν, τα που μπήκαν μνημόνια, όπως είναι η Κύπρος, αντιλαμβάνεστε. Και στην Κύπρο ειδικά ο αριθμός των εργαζομένων φτωχών, γιατί είναι αυτό το φαινόμενο που έχουμε τώρα, έχει υπερδιπλασιαστεί η κυβέρνηση λέει ότι μειώνεται η φτώχεια ή μειώνεται η ανεργία, αλλά όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουμε τους, είτε τους εργαζόμενους φτωχούς, είτε τους ανθρώπους που μεταναστεύουν, κυρίως τους νέους, για να μπορέσουν να βρουν κάπου αλλού στρίξη και βοήθεια και απασχόληση. Το ποσοστό της μερικής και προσωρινής απασχόλησης, χωρίς αυτό να είναι επιλογή των εργαζομένων, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και έχω αναφέρει τώρα μερικά από τα ποσοστά που οι πιο πολλοί το κάνουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή και είναι το ψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δραματική διεύρυνση της αγοράς υπηρεσιών και της ψευδοαπασχόλησης με πρωταθλητή το κράτος. Γιατί σήμερα πέραν του 30% των θέσεων στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα είναι θέσεις μη μόνιμες. Είναι ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου, αγορά υπηρεσιών και άλλα τέτοια για να γλιτώνει το κράτος από το να, προσφέρει μια εργασία με ασφάλεια. Επιπλέον έχουμε το κλείσιμο των κοινωνικών υποδομών, τα πάντα στον εθελοντικό τομέα. Περιμένουμε από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να λειτουργούν υπηαγωγεία, παιδοκομικούς σταθμούς, λέσχες ε, ε, για την απασχόληση των παιδιών. Τι εισηγούμαστε. Πρέπει να, που είναι βασική προϋπόθεση είναι η επαναρρύθμιση της εργασίας. Ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν όλους τους εργοδότες να εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις ε, εργασίας. Τη διασφάλιση ελάχιστων όρων απασχόλησης για όσους δεν καλύπτονται από τις συμβάσεις. Μέτρα που να αποτρέπουν την ψευδοαπασχόληση και να επαναφέρουν μισθούς και βελτίωση των όρων απασχόλησης και σίγουρα επαναδόμηση του κοινωνικού κράτους. Τι συζητείτε όμως σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα. Είναι το πακέτο Juncker, η πρόταση Juncker για τον κοινωνικό πυλώνα, που κατά εμά είναι γενικόλογες διακηρύξεις και δεν μπορούν να ανατρέψουν την νεοφιλελεύθερη ε, φιλοσοφία, το σύμφωνο σταθερότητα και άλλα. Εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο τι πολιτικέ τη ευελιξία, τη διαβίου μάθηση και την εθάριση τη κινητικότητα, με στόχο την εξυπηρέτηση του κεφαλαίου στην κατεύθυνση της εθάρρυνσης της κινητικότητας και η εισήγηση για δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Δεν συστήνουν βέβαια έναν όργανο που θα στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση και εργασία, αλλά περισσότερο για συντονισμό, ανταλλαγή απόψεων και πώ θα ε, εξυπηρετούν χωρί πραγματικά να δίνουν λύσει στο πρόβλημα τη απασχόληση και τη εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ξεπεράσατε κατά πάρα πολύ τον χρόνο που σας είχαμε δώσει, που ήταν δύο λεπτά. Ε, Εν πάση περιπτώσει όμως σας αφήσαμε να μιλήσετε γιατί τα είπατε τουλάχιστον πολύ ξεκάθαρα αυτά που θέλατε να πείτε. Ε, υπάρχουν μήπως ευρωβουλευτές που θέλουν ε, να πάρουν το λόγο, όχι από ό,τι φαίνεται. Δεν έχω κάποιον εγγεγραμμένο στον κατάλογό μου, λέει ο πρόεδρος. Αλλιώς ο κύριος Νικόλος ε, Μανιάς, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του, του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα του δώσω το λόγο λοιπόν. Ίσως θα συνεχίσει με στην ίδια γραμμή της προλαλής σας κυρίας, Ενδεχομένω. Θα το δούμε όμως. Ε, η γραμμή της ε, προηγούμενης ε, συναδέρφης και συντρόφισσας είναι μια ξεκάθαρα πολιτική γραμμή η οποία ε, εγώ θα πάρω πράγματα που, μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν τώρα. Αγαπητές ε, φίλοι και συνάδελφοι του Προεδρείου, Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, οι νέες μορφές εργασίας συχνά δεν προσφέρουν τα ίδια ωφέλη όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία με την εργασία πλήρους απασχόλησης και ενισχύουν το φαινόμενο της αδήλωτης και υποδηλωμένης, υποδηλωμένης εργασίας. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις νέες μορφές απασχόλησης με τη θέσπιση μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων με στόχο την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ειδικότερα ο στόχος των νομοθετικών ρυθμίσεων είναι να εμποδίσουν τη δημιουργία ανασφάλειας, να αντιμετωπίσουν την εφαρμογή των νόμιμων όρων εργασίας, να μειώσουν τις ανισότητες λόγω της σχέσης αυτής της ειδική σύμβασης και να εμποδίσουν την προσφυγή σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης για σκοπούς άλλους από εκείνους του οποίου έχουν νομοθετηθεί. Η πλήρη απασχόληση αποτελεί προτεραιότητα τη ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα για την άμεση υποστήριξη όσων των δυνατών περισσότερων ανέργων και την ένταξή του στην αγορά εργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική κυβέρνηση που ήταν τρία χρόνια, τέσσερα τα, τελευταία στο μνημόνιο με κυβέρνηση δική μας, μειώσαμε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες την ανεργία. Το 2018 το 72% της αύξησης των θέσεων εργασίας ήταν πλήρους απασχόλησης. Τον Αύγουστο του 2018 με την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών συμβάσεων και των διαπραγματεύσεων ευνοήθηκαν πάνω από 200.000 εργαζόμενοι. Θέλω μόνο μία παρατήρηση να κάνω, γιατί είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να πω, ότι η πολυμορφία και η πολυδιάσπαση των μορφών απασχόλησης που παρουσιάζονται εδώ και 20 χρόνια και ε, παραπάνω από 20 χρόνια είχαν εκφραστεί με την έννοια του απασχολήσιμου δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη συνοχή των δυνάμεων της εργασίας πράγμα που ανοίγει το δρόμο στις, στον δεξιό λαϊκισμό και στην ακροδεξιά. Γι' αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, της, αυτό, υπόψη μας να λάβουμε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, κύριε Μανιέ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Alice Μέρι Χίγκεν από την Ιρλανδία, που είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και είναι ανεξάρτητη. Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. Τώρα με ακούτε, πολύ ωραία. Στην Ιρλανδία αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι από αυτή τη συζήτηση για το επίπεδο της ανεργίας ένα επίπεδο ανεργίας το οποίο χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο με πολύ απλουστευτικό τρόπο Πηγαίνουμε τώρα, σιγά σιγά οδεύουμε προς μια κατάσταση στην οποία βιώνουμε κρίση από πλευράς ποιότητας απασχόλησης. Προς τα εκεί δηλαδή ε, κινούμαστε και είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Η έννοια ευελιξία ουσιαστικά έχει γίνει συνώνυμη της αβεβαιότητας, ενώ στην αρχή όταν το προέκυψε ο όρος ευελιξία ήταν κάτι που είχε να κάνει με την προβλεψιμότητα και το σχεδιασμό και την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής, προσωπικής και εργασιακής ζωής. Πρέπει δηλαδή να επανειδρύσουμε αυτή την έννοια, να έχουμε δομημένες ώρες, διαρθρωμένες, ποιοτική μερική απασχόληση, ακριβώς για να έχουμε ώρες στη διάθεση του εργαζομένου για την οικογενειακή προσωπική του ζωή. ευελιξία δηλαδή γι' αυτό ε, γεννήθηκε και ως όρος και ως ανάγκη και δεν θα πρέπει να είναι συνώνυμο της αβεβαιότητας. Επίσης πρέπει να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις για ατομικούς εργοδότες σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Έχουμε όλο και περισσότερους freelance, οι οποίοι είναι ψεύδο freelance. Υποτίθεται ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά τελικά δουλεύουν για ένα μόνο εργοδότη και είναι σαν υπάλληλοι και έτσι δεν έχουν κανένα χώρο για μια συλλογική διαπραγμάτευση, για να μπορέσουν να γίνουν τα δικαιώματά τους σεβαστά. Αυτό είναι πολύ δυστυχέ. Πρέπει να δώσουμε τον ορισμό του απασχολούμενου, του εργαζομένου. Ποιο είναι ο απασχολούμενος, ποιος είναι ο εργαζόμενος, τι σημαίνουν αυτοί οι όροι και ποιε είναι οι απώλειες για το κράτος από ε, τα έσοδα που δεν δηλώνονται από την αδήλωτη εργασία και ποιε είναι οι απώλειες για το άτομο και την προσωπική του ζωή όταν είναι αυτοαπασχολούμενο. Πρέπει να έχουμε λωρίδε απασχόλησης Δηλαδή, ε, λωρίδες εννοώ από πλευράς ε, οριαίου προγράμματος. Ε, δεν μπορεί κάποιος να, να μπορεί να το καλέσουν ανα πάσα ώρα και στιγμή. Θα πρέπει να μπορεί να απασχολείται εντός κάποιου συγκεκριμένου ωραρίου που μπορεί με ένα ποικίλει, αλλά να μην ξεπερνάει το ένα ανώτατο και κατώτατο όριο. Νομίζω ότι όντως ο νεοφιλελευθερισμός σπρώχνει το άτομο προς την αβεβαιότητα και τελικά ενισχύει τις κακές πρακτικές από πλευράς απασχόλησης. Χρειάζεται να εξετάσουμε το ζήτημα της εργασίας πρώτα ή της εκπαίδευσης πρώτα. για να προσαρμοστούμε στις νέες μορφές της απασχόλησης, τότε θα πρέπει η κατάρτιση να είναι ουσιαστική και αληθινή, να μην σπρώχνουμε το κόσμο σε βραχυπρόθεσμη εργασία ε, ε, αβέβαιη. Ήθελα να μιλήσω και για την ψηφιακή οικονομία. Νομίζω ότι η περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρξει ε, συνδικαλιστικό συνασπισμό σε μια ψηφιοποιημένη οικονομία, αλλά και η, περί, περίθαλψη είναι εξίσου σημαντική. Να έχουμε υψηλή ποιότητα απασχόλησης Υπάρχουν τομεί τη οικονομία όπου κυριαρχούν οι γυναίκε, όπω για παράδειγμα το τομέα τη περίθαλψη και των υπηρεσιών υγεία, που τελικά η, η κοινωνική φροντίδα σε αυτό το επίπεδο υστερεί σημαντικά. Και γίνεται και μία ανάθεση σε εξωτερικού αναδόχου, το outsourcing. Η δημόσια υπηρεσία ε, είναι δημόσια υπηρεσία, μπορεί να προσαρμοστεί στην καλή ποιότητα, μπορεί να καινοτομήσει, μπορεί να ανταλλάξει πρακτικές για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Επειδή όμως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες ε, αναθέτουν τόσο πολλά πράγματα σε εξωτερικούς αναδόχους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν καλύτερα. Και για τις κρατικές αγορές, τους δημόσιους διαγωνισμούς, πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρά μέτρα και να συζητηθεί αυτό το θέμα πραγματικά με ειλικρίνεια και σε βάθος. Ευχαριστώ. Ε, Uh, Ευχαριστώ. Έχουμε 10 λεπτά. Έχετε δυνατότητα να παρέμβετε και μετά. Επαναλαμβάνω το ερώτημά μου. Υπάρχει κάποιος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα θέλει να συμμετάσχει, να παρέμβει σε αυτό το σημείο στη συζήτηση. Έρχεται ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Τη Κοινοβουλής. Παρακαλώ, από τη Φιλανδία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Φιλανδός είμαι και το επίπεδο απασχόλησης ε, βελτιώνεται συνεχώς. Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο 6%. Παρ' όλα αυτά, έχουμε 200.000 ε, ελεύθερους επαγγελματίες, έχουμε όλο και πιο πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και είναι κάπως δύσκολη η κατάσταση, διότι μπορεί να είναι κανείς μερικός αυτοαπασχολούμενος, μετά να είναι άνεργος, μετά να είναι εργαζόμενος, μετά να είναι φοιτητής για ένα διάστημα και τέλος να είναι επιχειρηματίας. Και ο δημόσιος ε, τομέας, οι στατιστικές δυσκολεύονται να καθορίσουν τι ακριβώς ε, είναι ο άνθρωπος αυτός ε, και έτσι χάνει και τα ε, σχετικά επιδόματα ανεργίας. Προσπαθήσαμε να εισάγουμε ένα πρόγραμμα βασικού εισοδήματος, ελάχιστου εισοδήματος. Φαίνεται ότι υπήρχε ικανοποίηση, αλλά αυτό δεν δημιουργεί πολύ νέα απασχόληση. Προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους ε, να εργαστούν έστω και για σύντομα χρονικά διαστήματα. Τώρα όμως ε, δοκιμάζουμε μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Έχουμε ένα ψηφιακό σύστημα όπου μπορεί κανείς κάθε μέρα να εξετάζει τι δυνατότητες απασχόλησης υπάρχουν και αυτό συνδυάζεται με το επίδομα ανεργίας. Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν άλλες χώρες εδώ στην Ευρώπη που να έχουν ε, ανάλογα συστήματα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο νέο μοντέλο ελάχιστου εισοδήματος που να κινητοποιεί τους ανθρώπους περισσότερο από ό,τι τα καταφέραμε εμείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής από την Ρουμανία, η κυρία Τεβανδρέα Τσέρκε, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, κοινωνικών υποθέσεων ε, της Βουλής. Και εγώ θα μιλήσω τη χώρα της ε, χώρας μου, όχι τη μητρική μου. Θα μιλήσω στα ρουμάνικα πάντως. Νομίζω ότι είναι πολλές οι προκλήσεις στην αγορά εργασίας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που μπορούν να συμφιλιώσουν την επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά την απασχόληση, αλλά έχουμε και σοβαρά δημογραφικά προβλήματα. Σε μια γυράσκουσα Ευρώπη ε, υπάρχουν δύο λύσεις. Ε, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που συμφιλιώσουν βελτιώνουν και την ε, προσωπική ζωή και που δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες ε, και να είναι εργαζόμενες και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και έπειτα να δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να επανέρχονται στην αγορά εργασίας αρκετά γρήγορα, να έχουν τα κίνητρα έτσι ώστε να επιστρέψουν γρήγορα ε, στην αγορά εργασίας. Ε, στην Ρουμανία ε, προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά έχουμε και πολλούς πιο μεγάλους ανθρώπους, παπούδες που είναι ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται μη δραστήριοι ενώ θα έπρεπε ε, να μπορούν να εργάζονται ακόμα ε, και θα το ήθελαν και οι ίδιοι. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η ε, διαβίου κατάρτιση, να δούμε πώς μπορούμε σε όλους γίνεται περισσότερους ανθρώπους να αναπτύξουμε και τις ε, ψηφιακές ε, ικανότητες. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε το θέμα της ενεργούς ε, γύρανσης γιατί ε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν όλο και αργότερα ε, την δυνατότητα να ε, συνταξιοδοτηθούν, αλλά ακόμα και αν συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν δραστήριοι. Επίσης, η ενσωμάτωση των ανθρώπων με αναπηρία στην αγορά εργασίας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά η ασφάλεια των θέσεων εργασίας. Α, και βεβαίως πολύ σημαντικό και η ασφάλεια της εργασίας στο σπίτι. Θα πρέπει να καθοριστούν πολύ σωστά όλες ε, οι μορφές ε, εργασίας ε, και σε όλες τις μορφές αυτές να υπάρχει και η απαραίτητη ασφάλεια. Οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι καταρτήσεις στις ανάγκες αγοράς εργασίας και όχι μονάχα να μιλάμε για κατάρτιση για τους νέους ή για κάποιους νέους. Ε, να μιλάμε για καταρτήσεις οι οποίες ε, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και αίτημα των εργοδοτών, δηλαδή να μαθαίνουν δεξιότητες, να αποκτούν δεξιότητες που θα χρησιμοποιηθούν στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να τα βάλουμε στη φαρέτρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν την ε, διαδικασία. Θα ξαναδώσω όμως το λόγο στον Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα με προσοχή αυτά που υπόθηκαν και τρεις σύντομες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω σχετικά με έννοιες που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και που κατά τη γνώμη μου συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Πρώτον, ευελιξία. Κανείς ε, θα υποστήριζε ότι μπορεί ένας εργαζόμενος ε, να μην είναι ευέλικτος αλλά γιατί τι είδους ευελιξία μιλάμε, την ανεφόρον προσαρμογή του εργαζομένου όσον αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας, τον χρόνο εργασίας ή την ευελιξία να μπορεί να προσαρμοστεί σε νέες ε, μορφές και να μπορέσει να συμβάλλει στην παραγωγικότητα. Πολύ λίγο συζητιέται η μορφή της ευελιξίας και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά στο θέμα αυτό. Δεύτερον, χήμερα είναι το θέμα της ψηφιοποίησης. Γνωρίζω πολλούς που θεωρούν ε, την ψηφιοποίηση διαβολική κάτι πάρα πολύ κακό. Ενώ άλλοι θεωρούν ότι είναι αυτό που θα μας σώσει και που θα δημιουργήσει άπειρες θέσεις απασχόλησης. Εγώ έχω αμφιβολίες όσον αφορά το τελευταίο. Γνωρίζω από τις εργασίες της Επιτροπής μας εδώ στο Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν επιχειρήσεις σε μία που παράγει ξηράφια. Παλιά είχε 900 εργαζομένους. Τώρα έχει ψηφιοποιηθεί απολύτως και Σήμερα με τη διπλάσια παραγωγή έχει 9 απασχολούμενους. 9 εργαζόμενους. Όποιος λοιπόν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα ψηφιοποίηση και θέσεις απασχόλησης, θα πρέπει να το σκεφτεί. Θα πρέπει να σκεφτεί και την κατανομή της εργασίας. Να μην θεωρείτε όμως την ψηφιοποίηση την σωτηρία της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα, και στα κράτη-μέλη μας. Θα περιοριστώ σε αυτές τις δύο παρατηρήσεις. Ε, νομίζω όμως ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά όσον αφορά... να όσον αφορά το πώς ε, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την μελλοντική κατάσταση και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ε, επίσης, ε, δεν θα πρέπει απερισκεπτεί να σκεφτόμαστε θέματα όπως είναι το ελάχιστο ε, εισόδημα. Δηλαδή, το, η, η στάση πάρει αυτά τα χρήματα και ε, σταμάτα να παροπονιέσαι ε, δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε πιο ευφυή πρότυπα, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν με θάρρος και τόλμη να δημιουργήσουν νέες ε, συνθήκες απασχόλησης ε, και όχι να εμένουν σε πεπαλαιωμένες θέσεις. Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να νιώθουν δυσαρέσκεια όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης και την ε, αμοιβή που λαμβάνουν για την εργασία τους. Διότι έτσι θα απομακρύνονται από την κοινωνική Ευρώπη που θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε. Αυτά λοιπόν. Ε, νομίζω ότι σχεδόν εξαντλήσαμε το χρόνο μας. Ε, θα κλείσω εδώ και περνάμε ευχαριστώντας τον Άντριαν Σόλομον για την προεδρία του σε αυτό το πρώτο τμήμα της ε, συζήτησής μας. Ε, περνάμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης, το οποίο είναι εξίσου πολύπλοκο, εξίσου δύσκολο θέμα με το προηγούμενο. Okay. Ähm, wir steigen nun in den Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης συνεχιζόμενη εποπτεία και αξιολόγηση των δράσεων των κρατών μελών για άτομα με αναπηρία ως μόνιμο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχουμε και εδώ δύο βασικούς εισηγητές, ε, ομιλητές, ε, τους οποίους παρακαλούμε να μας κάνουν μια εισαγωγή στο θέμα αυτό. Την Κάρλα Ταβάρες, Μέλο τη επιτροπή ε, Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης ε, του Κοινοβουλίου τη Πορτογαλίας. Θα την παρακαλούσα να έρθει στο βήμα. Και δεύτερον, Άντε Μπάμπιτ, μέλος ε, της Επιτροπής Απασχόλησης Συνταξιωτικού Συστήματος και των Κοινωνικών Εταίρων του Κοινοβουλίου της Κροατίας. Σας παρακαλώ λοιπόν να έρθετε εδώ στο βήμα και έχετε ο καθένας πέντε λεπτά για την εισαγωγή σας. Παρακαλώ. So. Wer fängt an? Carla Tavares. Ja. Please. You have the floor. Bem, eu vou falar na minha língua materna, o português, pelo que peço-vos que coloquem já os escutadores para a tradução. Uh, e θα ήθελα να αξιοποιήσω την ευκαιρία που υπάρχει η για να μιλήσω στα πορτογαλικά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία θέλει να αποτελέσει ένα νέο υπόδειγμα για τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτό, σε αυτό το κλάδο. Επικυρώθηκε αυτή η σύμβαση στην Πορτογαλία και τα άτομα με αναπηρίες ήταν ε, μέρημνα από το 2009 που επικυρώθηκε αυτό το κείμενο όλων των πορτογαλικών κυβερνήσεων. Και με τον προπολογισμό του 2017 η κυβέρνηση αποφάσισε να παρέμβει σε αυτό το ε, πεδίο. Έτσι έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος για τη σχέση της κοινωνίας με αυτή την ομάδα πολιτών από πλευράς κυβέρνησης έχουν εφαρμοστεί διάφορα μέτρα και ενωτόμα για την καλύτερη συμπερίληψη και ένταξη στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες, με σεβασμό στην αυτονομία και στην ανεξαρτησία τους. Το μοντέλο στήριξης στην ανεξάρτητη ζωή είναι ένα από αυτά τα μέτρα. Τίθεται στη διάθεση αυτών των ατόμων μια ειδική υπηρεσία για να διενεργήσουν δραστηριότητε που ε, τους δυσκολεύουν από μόνοι τους, δεν μπορούν να τις κάνουν. Άλλο μέτρο είναι, είναι μοναδική κοινωνική παροχή για την κοινωνική προστασία των ατόμων, ενθαρρύνοντας την αυτονομία και την πλήρη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε. Το 2017 λοιπόν η κυβέρνηση προέβλεψε αυτό το επίδομα για την καταπολέμηση της φτώχειας και για να δώσει κίνητρο στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Απλουστεύεται το πλαίσιο των δικαιούχων και βελτιώνεται η κατάσταση. Το 2019 θα διευρυνθεί αυτό το μέτρο και θα συμπεριλάβουμε και τα παιδιά και τους νέους και θα ενισχύσουμε την κοινωνική προστασία νεότερων ατόμων και των οικογενειών τους. 88.000 άνθρωποι είναι δικαιούχοι αυτή τη στιγμή αυτής της ενίσχυσης, αυτής της παροχής και έτσι έχουμε περισσότερους πόρους για αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτή τη θητεία έχουμε εφαρμόσει και άλλα σημαντικά μέτρα όπως είναι η μείωση του φορολογικού βάρους για ε, το φορολογητέο εισόδημα από την εργασία των ατόμων με αναπηρίες φτάσαμε στο 14,5% την αξία των βοηθημάτων στο σπίτι και 3% για την ενίσχυση για την πληρωμή λογαριασμών. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής ε, των συμπολιτών μας και να έχουμε μια ολοκληρωμένη πανοπλία μέτρων για να λύσουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε και φοροαπαλλαγές, εξαιρέσεις από φόρους, πρόκειται για φορολογικό μέτρο με στόχο τη δυνατότητα να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να νοικιάσουν, να αγοράζουν οχήματα για να ε, κινούνται πιο εύκολα. και έχουμε και ε, ειδικέ πινακίδες κυκλοφορίας. Συνεργάζονται τα διάφορα αρμόδια υπουργεία με ένα πρόγραμμα πρόσβασης Plus, ΣΥΝ είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα με σειρά μέτρων για στήριξη των Δήμων, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των Δήμων, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χώρο και να προάγουμε την ισότητα μεταξύ των συμπολιτών μας. Και θέλουμε να περάσουμε στην ομοιόμορφη διαδικασία στο άειλο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας και δημόσιας διοίκησης για να έχουμε μια απολύτως ψηφιακή διαδικασία για όλα αυτά τα άτομα με αναπηρίες. Μη διάκριση των ατόμων στα project που συγχρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια. Αυτό είναι σημαντικό. Και Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί με φορολογικά πλεονεκτήματα. Έχουμε νέο ο καθεστώς εκπαιδευτικού συστήματος συμπερίληψης για όλους με μέτρα στήριξης στη μαθησιακή διαδικασία για να μπορούν όλοι οι μαθητές να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους. Και έχουμε ε, δουλειά στις σχολικές αίθουσες σε πολυτομεακό επίπεδο με τη συμβόλη των οικογενειών, των καθηγητών και των ειδικών υπευθύνων ειδική αγωγής και διαφόρων τεχνικών επαγγελμάτων. Με όλα αυτά θεωρούμε ότι έχουμε καταπολεμήσει την ανεπάρκεια και την, τον αποκλεισμό αυτών των ατόμων έτσι ώστε να είναι πλήρη και ενεργά μέλη στην κοινωνία μας. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την αυτοδιάθεση αυτών των πολιτών. Και τέλος, θέλω να υπογραμμίσω μια σειρά μέτρων της κυβέρνησής μας για την πρόσβαση στην απασχόληση. Για τη δική μας κυβέρνηση είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε μια στρατηγική πρόσβαση στην απασχόληση για όλους, και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα ε, στην Πορτογαλία. Έχει η κυβέρνηση οθετήσει μια στρατηγική προώθησης και προαγωγής της απασχόλησης με την ε, συμμετοχή διαφόρων φορέων, ε, διαφόρων δράσεων και στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην δυνατότητα μαθητείας και στάση της επιχειρήσης και σε ποσοστώσεις για αυτά τα άτομα με αναπηρίες που υποχρεωτικά πρέπει να τηρήσει ο ιδιωτικός τομέας. Και στις αρχές αυτού του μήνα άρχισε να ισχύει ένα νέο νομοσχέδιο, ένας νέος νόμος, ο οποίος υποχρεώνει τις εισηγμένες επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν με ποσόστοση άτομα με αναπηρίες, 1% ή 2% των εργαζομένων. Και θέλω να αναφερθώ στην έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών ε, της 6ης Φεβρουαρίου, έγκριση μιας σειράς μέτρων στήριξης στον άτυπο φροντιστή αυτών των ατόμων εντός της οικογένειας. Ε, είναι προτεραιότητα. Όλα αυτά είναι προτεραιότητα και είναι ένα υπόδειγμα, ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση για να βελτιώσει την αξιοπρέπεια ε, των ατόμων αυτών που αποτελούν μια πολύ ευπαθή κοινωνική ομάδα. Αυτά τα μέτρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, ε, μεταλαμπαδεύουν τις αξίες ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος για μια Ευρώπη πιο δίκαιη, πιο συμμετοχική, πιο δημοκρατική, πιο δίκαιη για όλους, όπου όλοι θα έχουν τη θέση τους, όπου κανείς δεν θα μένει πίσω. Αυτή την Ευρώπη ονειρευόμαστε, αυτή την ε, Ευρώπη επιθυμούμε και για αυτή την Ευρώπη θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και φτάνουμε στον επόμενο μιλητή, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ, όποιος θέλει το λόγο, έχουμε τώρα κίτρινα ε, έντυπα για όποιον θέλει να πάρει το λόγο, για να μην ε, μπερδέψουμε τις παρεμβάσεις. Ε, πολύ ευχαριστώ, λοιπόν. Θα λάβουμε το έντυπό σας. Δίνω το λόγο τώρα στην Άντε Μπάμπιτς, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Κροατικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε αυτήν την ε, ε, διακοινοβουλευτική ε, εβδομάδα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου γιατί διαπιστώνω ότι έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά με τους συναλλαγούς από τη Φιλανδία, από την Ρουμανία και προετοιμαζόμαστε ε, μάλιστα και για τις ε, ευθύνες μας ε, σε σχέση με το τρίγωνο συνεργασίας Φιλανδίας, Ρουμανίας, Κροατίας και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιπροσθέτως η συμπερίληψη ε, ανθρώπων που είτε έχουν αναπηρία είτε έχουν μειωμένη κινητικότητα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Η Κροατία ασκεί ε, τι, τους ε, μηχανισμούς σε πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής της ένταξης ε, στο στο, στην αγορά εργασίας. Ακολουθούμε τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών ε, για άτομα ε, με αναπηρίες καθώς επίσης ε, και σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική του 2010 και στην Κροατία έχουμε άλλωστε και εθνική στρατηγική. για την ε, συμπερίληψη ατόμων ε, με ε, αναπηρία. 78 καθορισμένα μέτρα από τα, τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε ήδη υλοποιήσει τα 43, για τα δε υπόλοιπα, από δε τα υπόλοιπα έχουμε 23 τα οποία είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο ε, και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και βεβαίως άρρηκτα συνδεδεμένο με το εξάμεινο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματο όλων των εκφάνσεων της, προσωπ... της επαγγελματικής κοινωνικής ζωής ε, σε ανθρώπους με αναπηρία. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατήσεις και μετά να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που ανέφερε ήδη η Πορτογαλίδα συνάδελφος όσον αφορά την κοινωνική προστασία ε, και όσον αφορά την προσβασιμότητα των υπηρεσιών ε, για παιδιά τα οποία είτε πάσχουν από φυσική είτε από πνευματική αναπηρία ή στέρηση ανάπτυξης επίσης ε, επιδόματα έτσι ώστε ε, η υλική κατάσταση των αναπήρων να βελτιωθεί. Βελτίωση της ε, προσβασιμότητας στην απασχόληση. Ποσοστώσεις έχουν σημειωθεί και έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και συστηματικά ε, δίνεται η δυνατότητα για βοηθό της σχολικής ε, ζωής στις περισσότερες ε, περιπτώσεις. Επίσης, λαμβάνονται μέτρα τα οποία αφορούν την βελτίωση των συνδικών εργασίας και της απασχολησιμότητας ε, των ε, ανθρώπων με αναπηρία. Ε, αυτό το μέτρο θα πρέπει να δείξει σύν το χρόνο εάν είναι ικανοποιητικό. Επίσης, η αποϊδρυματοποίηση κυρίως νέων ανθρώπων ε, που αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι στην δημοκρατία της Κροατίας παρότι έχουν ε, ληφθεί πολλά μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και επαγγέλματο για τα άτομα με αναπηρία παρόλα αυτά ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο το επιθυμητό. 70.000 ε, άνθρωποι ε, που θα μπορούσαν με κάποιες προσαρμογές ε, να βρουν θέση απασχόλησης μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέσα μεταφοράς γιατί αυτά δεν είναι πάντα προσβάσιμα και δεν έχουν τη δυνατότητα ε, προσαρμογής ε, της ε, κατοικίας έτσι ώστε η, να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους. Επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι ακόμα δεν έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους και μηχανισμοί που ακόμα δεν έχουν καν εφαρμοστεί. Θα πρέπει επομένως να καταβληθούν πολύ περισσότερες προσπάθειες έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να παραμείνουν στην οικογένειά τους, να διατηρήσουν το μέγιστο βαθμό ε, ε, ανεξαρτησίας ε, και να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στα σπίτια τους. Θα πρέπει, δεν άκουσα τη συνάδελφο Ταβάρες να αναφέρεται σε αυτό, θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία οποιοδήποτε είδους να μην ιδραματοποιούνται. Ε, εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από ιδρυματοποίησης, ίσως όμως με λάθος τρόπο, γιατί ε, άτομα με βαριά, με βαριές αναπηρίες ε, έχουν βγει από τα ιδρύματα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν, να προκληθούν και άλλα προβλήματα. Ε, προβλήματα. Επομένως θα πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις προσπάθειες που κάνουμε την 1η Ιανουαρίου του 2019 πέρασε ένας νέος νόμος ε, για την εντατικοποίηση της αποϊδρυματοποίησης έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μην μπαίνουν ε, στα ιδρύματα και να μην κλείνονται σε αυτά αλλά να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ε, στα, πατρικά του σπίτια έχοντας βέβαια και τη δυνατότητα για βοήθεια στο σπίτι. Προσπαθούμε λοιπόν να δουλέψουμε σε τρία επίπεδα. Ε, σε, στο επίπεδο αυτής της ε, βοήθειας ή του βοηθού ε, στο σπίτι, στο επίπεδο της φυσικοθεραπείας και της ιατρικής φροντίδας και βεβαίως της δυνατότητας παροχής οδηγίας σε περίπτωση που η αναπηρία δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα. Όλοι θέλουμε ε, θετική Ευρωπαϊκή Ένωση και μια Ένωση Ευρωπαϊκή η οποία θα ακτινοβολήσει παγκόσμιο επίπεδο όχι μόνο οικονομικά αλλά και για λόγους δημοκρατίας αλλά και για λόγους προστασίας των πιο ευάλωτων τμήματων του πληθυσμού. Αν θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να πετύχουμε ένα τέτοιο στόχο, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη θέση των πιο ευάλωτων ομάδων ε, στις, ε, ε, στους πολίτες μας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στο Κροατικό Κοινοβούλιο, σε αυτήν την θητεία καταφέραμε κάτι θετικό, να δώσουμε βήμα ε, σε ε, άτομα με αναπηρία και σε άτομα τα οποία κυκλοφορούν με αναπηρικό αμαξίδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουν ζητήσει διάφοροι το λόγο. Ε, και εάν θέλει κανείς άλλο το λόγο, σας παρακαλώ να τον ζητήσει μέσα στα επόμενα λεπτά, διότι σύντομα θα κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών για να ολοκληρώσουμε εν καιρό στη συζήτηση. Σβετλάνα Αγγέλοβα, παρακαλώ. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, в рамките Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συνεχίζουμε τη δουλειά μας για να ενθαρρύνουμε τη συμπερίληψη στον εργασιακό ιστό των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των ατόμων με αναπηρίες. Ε, έγινε μια ψηφοφορία τον περασμένο Δεκέμβριο και θέλω να σας ευχαριστήσω την προσοχή σε αυτή την ε, ψηφοφορία για τα άτομα με αναπηρίες και εφαρμόσαμε μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματος της κυβέρνησής μας. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν για την εγγύηση των θέσεων απασχόλησης των ατόμων που παρουσιάζουν κάποια αναπηρία σε ε, ειδικό και προστατευμένο περιβάλλον. Υπάρχει νόμος που προβλέπει τη χορήγηση επαρκούς στήριξης για τα άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται αλλά και για τον εργοδότη τους. Ο νόμος λοιπόν προβλέπει προς ποσοστώσεις για το εργασιακό δυναμικό για να ενισχυθεί η απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες στο συνήθι χώρο εργασίας για να μπορούν να έχουν και έσοδα από τη δραστηριότητά τους. Έχουμε φτιάξει ένα ειδικό ταμείο για την απασχόληση για τα άτομα αυτά. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής προβλέπει να θεσπίσει και να υλοποιήσει ειδικά προγράμματα για να ενθαρρύνει την απασχόληση και για να ενθαρρύνει τους εργοδότες να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης που θα απευθύνονται σε άτομα με ε, ε, βιώσιμη αναπηρία. Έχουμε κέντρα απασχόλησης, είναι μηχανισμοί ένταξης στην αγορά εργασίας και όλα αυτά τα κάνουμε επειδή έχουμε ψηφίσει το συγκεκριμένο νόμο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Έχουμε βελτιώσει την πρόσβαση στην απασχόληση και στην κατάρτιση για να βελτιωθούν και τα επαγγελματικά προσόντα και να βελτιωθούν και τα εργασιακά προσόντα των ε, ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Στην ώρα σας ολοκληρώσατε. Ο κύριος Νίκολας Μανιός, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Η ελληνική κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στην κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη. Υγειάται τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες στους βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως στην παιδεία με τη διεύρυνση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και των τμήματων ένταξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την αύξηση του αριθμού των προλήψεων προσωπικού και των διορισμών για πρώτη φορά εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή με την ενίσχυση της προσβασιμότητας των σχολικών κτηρίων με την κάλυψη για πρώτη φορά μαθητών που χρήζουν παράλληλη στήριξη. Στην κοινωνική πολιτική με την ψήφιση του νόμου υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται πλέον ως ισότιμη με την ελληνική και την ελληνική και την ελληνική γραφή Μπράιλ να αναγνωρίζεται ως ο τρόπος γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών με τη δράση δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για την αυτόνομη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη θάλασσα με την καθιέρωση του 15% των προλήψεων στο δημόσιο να καλύπτεται από άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους με τη δημιουργία σημείων αναφοράς σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια της χώρας για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ. Μέτρα κοινωνικής φροντίδα, με τον νόμο και την αναδοχή και την υιοθεσία με στόχο να μην μένει κανένα παιδί στα ιδρύματα με το πιλωτικό πρόγραμμα αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία και μεταστέγαση σε δομές φιλοξενίας με τον ηλεκτρονικό γενικό εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ατόμων με αναπηρία με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία για την ένταξη ευάλωτων ειδικών ομάδων στην αγορά εργασίας με στέγες υποστηριζόμενες διαβίσεις, τις κατασκηνώσεις για όλους, την ισότιμη πρόσβαση στον ΑΜΕΑ, στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Ακόμη έγιναν προσπάθειες από την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια όσο διαρκούσε το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής να μην κοπεί ούτε ένα ευρώ από τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία. Το ποσό που καταβάλλεται ως προνοιακή παροχή στα άτομα αυτά δεν φορολογείται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο. Ιδιώτε ή πιστοτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται τα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Άνταμ Κρούζερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ. Είναι αργά. Ε, χαίρομαι που άκουσα όσου πήραν το λόγο. Εδώ και 10 χρόνια είμαι ευρωβουλευτής. Από την Ουγγαρία προέρχομαι. Είμαι κοφός. Ειδικεύομαι στο θέμα των ίσων ευκαιριών και εκπαίδευση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, η απασχόληση των ε, ατόμων με αναπηρίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται γύρω στο 50%. Στην Ουγγαρία είχαμε το 20% το 2011, τώρα έχουμε βελτιωθεί, έχουμε ποσοστό 40%, αλλά βέβαια το ποσοστό κυμαίνεται ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους δύο προλαλήσαντες που μίλησαν για μέτρα που απαιτούνται για να αλλάξει η κατάσταση. Δεν θέλω να σας απαριθμίσω όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, ε, ούτε όλα τα μέτρα που έχουν αναλυφθεί στην Ουγγαρία ή σε άλλες χώρες. Θα ήθελα να περιοριστώ σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η κατάσταση στην αγορά εργασίας πρέπει συνεχώς να αξιολογείται με στόχο την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρακτικές που αντίκυνται στην απασχόληση ατόμων με αναπηρίες. Τρίτον, θα πρέπει να έχουμε ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας, ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Επίσης, ε, εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντικά θέματα, όχι μόνο για άτομα με αναπηρίες, αλλά για όλους και για τους εργοδότες. Συχνά οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αρκετά ο ένας για τον άλλον. Είναι πολύ σημαντική και η διαβίου εκμάθηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην δέσμη μέτρων για την προσβασιμότητα που υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο του χρόνου. Θα πρόκειται για υποχρεωτικά μέτρα, δεσμευτικά για όλα τα κράτη-μέλη και ελπίζω έτσι να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την προσβασιμότητα. Ελπίζω η σημερινή συζήτηση επίσης να φανεί χρήσιμη. Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ο ένας τις βέλτιστες πρακτικές του άλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η άλλη Μέρι Χίγγιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να φέρω ε, ένα-δύο πράγματα. Ξέρω ότι μακρηγόρησα πριν. Κάτι που κάναμε πρόσφατα στην Επιτροπή Κοινωνικής προστασία ήταν να προσπαθήσουμε να έχουμε κοινέ συνεδριάσεις με την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή Εκπαίδευσης στο Κοινοβουλίο μα ιδιαίτερα για το θέμα των ατόμων με αναπηρία. Ε, διότι διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διάφορε σειρέ κανόνων και πολλή γραφειοκρατία. Υπάρχει δηλαδή πολλή δουλειά στην διαχείριση μιας αναπηρίας. Πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς τη γραφειοκρατία ενός συστήματος υγείας, ή όταν μεταβαίνει κανείς από ε, ένα σύστημα εκπαίδευσης σε ένα σύστημα απασχόλησης, βλέπουμε πάλι γραφειοκρατία που μπορεί να εμποδίσει την πρόοδο. Έχουμε κάποια θετικά σημάδια στην ε, Ιρλανδία, έχουμε κάποια μέτρα ε, σωστής προσαρμογής στον χώρο εργασίας, κάτι που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη στιγμή. Δυστυχώ όμως τα διάφορα συστήματα που εφαρμόζονται συχνά δεν συνδυάζονται πολύ καλά μεταξύ τους. Πέρα από την πρόσβαση στον χώρο εργασίας, ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία συζήτηση σχετικά με την πρόοδο των ε, ατόμων αυτών, τη σταδιοδρομία του. Δηλαδή να μην βλέπουμε την απασχόλησή του ω μία κατάσταση, πρέπει να βλέπουμε και τη δυναμική πορεία τη σταδιοδρομία του. Ε, θέλουμε να δούμε τέτοια άτομα και στα διοικητικά συμβούλια ε, ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις στην κορυφή των ε, διαφόρων φορέων. Επίσης, όσον αφορά το πρωτόκολλο ε, θα ήθελα να ρωτήσω, επικυρώθηκε το ε, προαιρετικό πρωτόκολλο της ε, σύμβασης του ΟΗΕ. Πολλοί από τους κοινωνικούς στόχους αναφέρονται ως ποσοστό σύγκρισης με άλλες χώρες. Πώς λοιπόν μπορούμε να έχουμε ποιοτικού δείκτες στην ε, διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, ε, μια νότα ανησυχίας ακόμα και πέρσι. Ε, μας είπαν ότι η Ιρλανδία δαπανεί πολλά στο σύστημα υγείας. Πώς λοιπόν μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο ένα μήνυμα και στο άλλο. Δηλαδή ότι δαπανούμε ε, πολλά χρήματα, από την άλλη έχουμε ανθρώπους που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους ε, σύμφωνα με ε, την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν θα δυσκολευτώ διότι έχω την κυρία Σκέβη Κούτρα Κουκούμα, μάλλον λάθος προέβρα το όνομα, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. Πρόεδρε, να πω ότι ως Κύπρος έχουμε κυρώσει από το 2011 την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Είχαμε κάνει μια πρώτη, ε, ένα πρώτο σχέδιο δράσης ε, από το 2013 μέχρι το 2015. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν η περίοδος της κρίσης και έτσι πολύ λίγα πράγματα είχα γίνει. Βέβαια υπάρχουν οι στοχευμένες πολιτικές τις οποίες συζητούμε πολύ συχνά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναδεικνύονται τα κενά και οι αδυναμίες που μπορεί να διαμορφώνουμε ωραιότατες στρατηγικές και σχέδια δράσης για τα οποία αν δεν ξεπεραστούν η γραφειοκρατία και αν δεν ε, δεσμευτούν κονδύλια αντιλαμβάνεστε θα μείνουν στο χαρτί ως ωραίες στρατηγικές. Η τελευταία στρατηγική 1828 που έχει διαμορφωθεί βασίζεται και στις παρατηρήσεις που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν υποδείξει στην Κύπρο όπως και στην Ευρωπαϊκή, ε, από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και την Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εμείς θεωρούμε, μέσα από τη συζήτηση σήμερα έχω ακούσει και πολιτικές και σχέδια που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες που ενδεχομένω όπως έχω ακούσει, πολύ πιο προχωρημένα που εμείς θεωρούσαμε ότι είχαμε πολύ ε, σωστά, όπως είναι η ποσόστοση της προσλήψης ε, στο δημόσιο τομέα, όπου για μας ήταν μόνο 10% και αντιλαμβάνεστε λόγω της οικονομικής κρίσης και του memorandum στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, δεν έχει προσληφθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια σχεδόν κανένας. Τώρα ενδεχομένως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, επίσης, μέσα από το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, όπου έχουν μπει κάτω και τα άτομα με αναπηρία, υπάρχει μεγάλη αδικία σε βάρος τους και είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε με ποιον τρόπο να ξεπεράσουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε είναι θέμα της κυβέρνησης. Ε, όπως και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι ανάγκη να αναλύσω, για μας είναι πολύ σημαντικό α, η παρακολούθηση και ο έλεγχος τον, το ότι έχει σκυρώσει μια σύμβαση να μην είναι μόνο στο χαρτί όπως έχω πει στην αρχή και να πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την οργάνωση των ατόμων με αναπηρία όπου έχουν έτσι πολύ καλές τοποθετήσεις σε σχέση με το πώς πραγματικά εφαρμόζεται και δεν υπάρχει η, η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και πραγματικά δεν υπάρχει καμιά διάκριση σε βάρος των ατόμων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κωνσταντίν Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που ακούω για τις θετικέ εξελίξεις στις πιο φτωχέ χώρες του Νότου, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Επειδή είναι σημαντικό να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχει σημασία να τονίσουμε πως στις χώρες αυτές, αν και υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, οι αριστερές κυβερνήσεις επιλέγουν να κάνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους με αναπηρία. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα για τη χρηματοδότηση της βοήθειας στο σπίτι, γιατί είναι μια από τις προτάσεις που έχω κάνει για το οικιακό προσωπικό και τους φροντιστές η δυνατότητα παροχής βοήθειας στο σπίτι είναι πολύ σημαντική για τους ανάπηρους και μεγάλη ανακούφιση για τις οικογένειες που δεν έχουν πάντα την εξειδικευμένη γνώση που χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει πολλή δουλειά σε αυτά τα θέματα, αλλά συχνά συναντούμε δυσκολίες στο Συμβούλιο. Άρα η συνεργασία μαζί σας για να ασκείτε πίεση τη κυβερνήσει σα είναι απαραίτητη και πολύτιμη. Έχουμε ζητήσει, για παράδειγμα, προγράμματα που βοηθούν στην προσαρμογή στην εργασία και στο περιβάλλον των σπιτιών. Οι κυβερνήσει θεωρούν πολλέ φορές τέτοια προγράμματα ω πολυτέλεια. Σα διαβεβαιώνω πω δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασική ανάγκη αυτονομία που μα είναι πολύτιμη. Και θα ήθελα να, να πάω και ένα βήμα πέρα από αυτό. Χρειάζονται όλοι μαθήματα συμβίωσης με ανθρώπους με αναπηρία. Οι συνάδελφοι στη δουλειά, η συνύπαρξη στο σπίτι, να βοηθήσει όλους και θα δώσει στους ανθρώπους χωρίς αναπηρία την εδότητα να καταλάβουν τι βιώνουμε. Κάτι τέτοιο νομίζω μας κάνει όλους καλύτερους ανθρώπους. Επίσης, όταν μια χώρα δίνει ε, βοήθεια στο σπίτι, μια κυβέρνηση δίνει βοήθεια στο σπίτι, Οπωσδήποτε πρέπει να έχει και εκπαίδευση για το οικιακό προσωπικό. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε κινητικότητα οικιακό προσωπικό. Γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε ένα άνθρωπο χωρί να έχει κάνει κατάρτιση, χωρί να έχει πιστοποίηση στο επάγγελμα, να πληρώνεται από πόρου, από προγράμματα το κράτος και να το στέλνουμε στα σπίτια, γιατί μπορεί να μην πετύχουμε το στόχο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Τότε οπωσδήποτε αναγνώριση και πιστοποίηση του επαγγέλματος. Χωρίς αυτό δεν θα κάνουμε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφο Ντεμπατούλ έχει το λόγο, παρακαλώ. Αν βλέπω καλά, λέει ο πρόεδρος από το Βέλγιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κείμενο που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο των Βρυξελών που λέει ότι οι τοπικές διοικήσεις θα πρέπει να έχουν στο προσωπικό τους 2,5% άτομα με αναπηρία αυτή η υποχρέωση ε, προκαλεί προβλήματα ε, και διευρύναμε λοιπόν το μέτρο αυτό ε, λέγοντας ότι αυτή την υποχρέωση θα μπορούσαμε να τη δώσουμε κατά κάποιο τρόπο σε υπεργολαβία περνώντας αυτή το μισό της υποχρεωμένης, ε, υποχρεωτικής συγγνώμη, ε, ε, μέσα από διαγωνισμούς και διαδικασίες ανάθεσης σε πιο εξειδικευμένες εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στην τοπική διοίκηση να σεβαστεί το νόμο, γιατί ναι μεν εφήρμοσε τον νόμο αλλά προώθησε εργαζόμενους σε άλλες ε, μορφές γιατί και με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στους ε, ε, ανθρώπους με αναπηρία να εργαστούν αλλά δόθηκε και η δυνατότητα και στις τοπικές διοικήσεις να έχουν στα πλαίσια τους ανθρώπους με αναπηρία αλλά και να απομυθοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο και εντό εισαγωγικών την σχέση με ανθρώπους με αναπηρία. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι υπήρξε και η απαραίτητη παρακολούθηση. Επίσης η εμπειρία καταδεικνύει ότι στις τοπικές αρχές, στην δημόσια διοίκηση και στον πρώτο βαθμό της διοίκησης διαπιστώνουμε ότι το γεγονός ε, της ύπαρξης ε, ε, ανθρώπων με αναπηρία στα πλαίσια του προσωπικού ε, είναι πολύ θετικό και επίσης ε, ακόμα και οικονομικά αποδοτικό γιατί πρόκειται για προσωπικό το οποίο απουσιάζει σπάνια και το οποίο δουλεύει πολύ καλά και επομένως πραγματικά προσυπογράφω και σημειώνω την ανάγκη να υπάρχουν άτομα με αναπηρία στο προσωπικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ράφκα Μάξοβα είναι η τελευταία ομιλήτρια. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι που συζητάμε εδώ το θέμα των ανθρώπων με αναπηρία. Στην Σλοβακία έχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας, ωστόσο υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Περίπου πριν δύο χρόνια δημιουργήσαμε ένα όργανο εποπτείας για τα άτομα με αναπηρίας και πιστεύουμε ότι έτσι θα έχουν καλύτερη θέση τα άτομα αυτά όσον αφορά τις ε, κοινωνικές παροχές. Ελπίζουμε ότι θα ενταχθούν καλύτερα στην κοινωνία τα άτομα αυτά. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να ενταχθούν καλύτερα στην κανονική ζωή και να μην αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών από το κράτος και για τους εργοδότες ε, οι οποίοι εάν ε, προσλάβουν αρκετά άτομα με αναπηρίες ε, έχουν κάποια πλεονεκτήματα. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορούν να προσλάβουν άτομα με αναπηρίες, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν ε, τέτοια άτομα και αν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, τότε πληρώνουν ε, κάποιο τέλος στο κράτος. Ένα φαινόμενο που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη είναι αυξανόμενος αριθμός ψυχικά ασθενών ε, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι τάση αυτή πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει. Ε, μπορούμε όμως να έχουμε μοιρασμένες θέσεις εργασίας και καλύτερη κοινωνική προστασία. Θέλουμε να έχουμε υπηρεσίες ανακούφισης των ανθρώπων αυτών, κοινωνική νομοθεσία και τα άτομα με σημαντικό βαθμό αναπηρίας ε, λαμβάνουν ε, ε, επίδομα από το κράτος. ...6,8 δισεκατομμύρια επενδύσαμε πέρσι στα άτομα με αναπηρίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Πρέπει να ομολογήσω ότι ως άτομα χωρίς αναπηρία η σημερινή συζήτηση ήταν ε, σαν η μερίδα βέλτιστων πρακτικών. Ακούσαμε τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη. Ήμουνα παλαιότερα σε Διοικητικό Συμβούλιο Επιχείρησης και είχαμε μια ειδική εκδήλωση για άτομα με βαριά αναπηρία, όπου είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν, αλλά δεν υπήρχε σχεδόν κανένας τρόπος ανταλλαγής ε, απόψεων ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα χωρίς αναπηρία. Ίσως εκεί να βρίσκεται το κλειδί, η λύση. Διότι νομίζω ότι τα άτομα χωρίς αναπηρίες ασχολούνται πολύ λίγο με το θέμα αυτό. Με το πώς δηλαδή μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει και εγώ να προβληματιστώ περισσότερο πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως απλά στο τέλος αυτής της συζήτησης να εκφράσω τη σκέψη αυτή για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ε, ο Άνταμ Κόζα, η Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης που ασχολούνται με το θέμα των ανθρώπων με αναπηρία. Και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα συνεχίσουμε και τις επαφές με τις ανάλογες επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Θα σας παρακαλούσα ή μάλλον να σας θυμίσω ότι θα περάσουμε τώρα για το γεύμα στο σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Παρακαλώ μην αφήσετε προσωπικά σας αντικείμενα εδώ στο, στην αίθουσα, διότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ξαναμπείτε στην αίθουσα για να τα πάρετε. Σας παρακαλώ λοιπόν να πάρετε όλα τα προσωπικά σας αντικείμενα μαζί σας. Άντριαν Σόλομον. Αχ, σας ξέχασα, συγγνώμη. Ε, ladies and gentlemen, moment, please. Καθίστε λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, γιατί συμμετείχατε σε αυτήν την διακοινοβουλευτική διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο υπό την Προεδρία της Ρουμανίας. Να προσθέσω ότι τα δύο θέματα του σημερινού μας πάνελ ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικά, αλλά παρουσιάζουν και κοινά στοιχεία. Ε, η ψηφιοποίηση, ε, η συμπερίληψη ανθρώπων με αναπηρία, αυτά μας οδηγούν στην ανάγκη κοινής δράσης. Η τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες και που ε, γίνεται όλο και πιο απτή γύρω μας κάθε μέρα, μπορεί ας πούμε να βοηθήσει όσους έχουν προβλήματα όρασης. πλάστικ Astăzi γιατί διαφορετικά, ε, ε, ε, συγγνώμη, παλιότερα οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δούλευαν σε κάποιες θέσεις πολύ χαμηλού επίπεδου, ενώ τώρα στη Ρουμανία έχουμε τυφλούς εργαζόμενους που χρησιμοποιούν τη μέθοδο Μπράγ και που δουλεύουν σε συστήματα πληροφορικής κλπ. Επίσης, στην ε, Ρουμανική Γερουσία έχουμε ένα σχέδιο δράσης ε, που αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών στην Ρουμανία έχουμε περίπου 800.000 ανθρώπους με αναπηρία. Οι περισσότεροι από αυτές τις 800.000 παίρνουν διάφορα ε, επιδόματα, βοηθήματα, έτσι ώστε να μην βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά αντιθέτως ε, να συμπεριληφθούν κοινωνικά στην ε, ζωή και στην καθημερινότητά τους μέσα από βοήθεια στο σπίτι κλπ. Είναι γεγονός όμως ότι πρέπει να ε, υπάρξει και η συνεργασία με το τοπικό επίπεδο γιατί στα, στα δημαρχία, στα ε, διοικητήρια, στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν ακόμα όλες ε, οι δυνατότητες που πρέπει να υπάρχουν όπως ας πούμε για τη βοήθεια ανθρώπων τυφλών ή για κοφαλάλων με την νοηματική γλώσσα. Γι' αυτό είναι σημαντικό με ε, χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία να ε, καταρτιστούν οι υπάλληλοι, η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών που εργάζονται με άτομα με αναπηρία. πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι άνθρωποι με αναπηρία θα έχουν την δυνατότητα και πρέπει να έχουν την δυνατότητα να εντάσσονται στην κοινωνία, να έχουν πρόσβαση ε, στα μέσα μεταφοράς, να έχουν πρόσβαση στην κινητικότητα και επομένως να έχουν ανοιχτές όλες τις δυνατότητες που δίνει η κοινωνική ζωή και φυσικά την ε, ε, δυνατότητα να χρησιμοποι... να ε, ε, ζουν με ανεξαρτησία τη ζωή τους όπως ακριβώς το επιθυμούν. Η εντυπωσία είναι πιο active, da Επίσης θα πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα σε άτομα ειδικά με αναπηρία, ε, η δυνατότητα λέω της τηλεεργασίας, δυνατότητα δηλαδή να εργάζονται από το σπίτι τους έτσι ώστε να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, έτσι ώστε να ε, σταματήσουν να θεωρούνται πάντοτε ε, άτομα έθραυστα και τροτά. Οι στόχοι λοιπόν είναι σωστοί, ε, αλλά θα πρέπει να ενταχθούν στους στρατηγικούς στόχους και τις δημόσιες πολιτικές. Ωραία λοιπόν, ολοκληρώσαμε για τώρα, θα τα πούμε αργότερα στο δείπνο. Ελπίζω να σας ε, άρεσε αυτός ο ε, επικοδομητικός διάλογος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σα ευχαριστώ πολύ και πάλι, Άντριαν, σου ζητώ συγγνώμη για το λάθο μου.